η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθήσουμε δηλαδή οικολογικές, οικολογικές πράσινες μορφές διαβίωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι ε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού που είναι άνω των 50 και ένα άλλο ποσοστό το οποίο θα θέλει να φτάσει προφανώς στα 50 σε καθεστώς πλήρους υγείας. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε πιο οικολογικούς πράσινους τρόπους διαβίωσης, μήπως θα πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερο λαχανικά και λιγότερο κρέας, μήπως θα πρέπει να έχουμε πιο οικολογικούς τρόπους μετάβασης στις δουλειές μας για παράδειγμα θα θέταμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πολύ θετικό παράδειγμα, να το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα μπορούσε να διασφαλίσει ότι τέτοιες συνεδριάσεις θα γίνονται στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο. Κύριε Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπη, σίγουρα η ενεργειακή μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία είναι θεάριστος στόχος και χαίρομαι γιατί αποκαλέσατε το Ταμείο, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Βέβαια είναι κάπως γενική και όριστη προς το παρόν η πρόταση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι λεπτομέρειες. Ελπίζω στην πορεία να τα διευκρινίσετε καλύτερα αυτά, κύριε Τίμερμανς. Γιατί για το επενδυτικό σχέδιο του πρώην Πρόεδρου Γιούνκερ, Δυστυχώ τα κονδύλια επικεντρώθηκαν σε ορισμένε χώρε μόνο. Φυσικά και χρειαζόμαστε επενδύσει και μάλιστα επενδύσει σε πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Αυτές τις επενδύσεις ε, ε, και αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε και άλλους τομείς να υλοποιήσουν την απαλλαγή τους από τις εκπομπές άνθρακα και να δούμε φυσικά και τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες και να λάβουμε υπόψη τις ειδικέ ανάγκες της κάθε χώρα και του ενεργειακού, των ενεργειακών του μειγμάτων. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής ε, του Προέδρου. Πάνω από 50 ε, πρωτοβουλίες ε, της Κομισιόν ε, αναμένουμε Οπότε σίγουρα ε, σε κάθε ε, ολομέλεια θα έχουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα, οπότε θα καλυφθούν φαντάζομαι οι, ε, όλες οι πτυχές και θα ακουστούν όλες οι απόψεις. Έτσι για να κλείσει η συζήτηση αυτή τη φορά θα ήθελα να δώσω για μια ακόμη φορά στους δύο αντιπροέδρους και πρώτο το λόγο έχει ο κύριος Τίμπερ. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Εάν δεν περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου, δεν θα ελέγχουμε πλέον το πεπρωμένο μας, τη μοίρα μας. Θα βγουν εκτός ελέγχου τα πράγματα, ε, θα είναι πάρα πολύ καταστροφικά τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν δεν μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θα το κάνουν άλλοι αντί για εμάς. Και εγώ πιστεύω ότι κάποιοι θα βγουν πολύ κερδισμένοι, αλλά είναι και πολλοί αυτοί που θα χάσουν. Και αυτό είναι το μήνυμα. Ε, και με την προειδοποίηση τι κάνει κανείς, Είδε την αγνοή και συνεχίζει ε, σαν να μην τρέχει τίποτα, όπως κάποιοι φαίνεται να ε, υποστήριζαν, μπορεί κάποιος να κρυφτεί και να χωθεί κάτω από το κρεβάτι ή να αρχίσει να δρά. Και αυτό κάνουμε εμείς. Αυτό κάνουμε στην Κομισιόν με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Κάποιοι λέτε δεν αρκεί. Όχι, δεν αρκεί. Έχετε δίκιο. Θα χρειαστούν περισσότερες προσπάθειες. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και όλα τα ταξίδια έτσι ξεκινάνε με ένα πρώτο βήμα. Και θα αρχίσουμε να συζητούμε μαζί σα τα διάφορα στοιχεία στου επόμενου μήνε, τα επόμενα χρόνια, για να το πετύχουμε. Και θέλω να ευχαριστήσω όλο ιδιαίτερος ε, τον πρόεδρο Μπούζεκ, ο οποίο κατέθεσε την πρόταση αυτή, γιατί δική του ιδέα είναι και εμείς αυτή την ιδέα επεξεργαστήκαμε. Και θα ήθελα αυτή την ημέρα να το πω. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από ακριβώ ένα χρόνο ένας δήμαρχος, ο Πάβελ Αντάμοβιτς, πολύ θαραλέος δήμαρχος και φίλος μου, δολοφονήθηκε. Ο Πάβελ ήταν υπέρ του διαλόγου ε, και της ε, ελευθερίας. Ήθελα να αναφέρω το όνομά του σήμερα, να τον μνημονεύσω γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ε, και να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και θα πω ναι, πράγματι είμαι ε, και εγώ εγγονός ε, ανθρακορίχων. Γνωρίζω όμως ότι έχει χτυπήσει το καμπανάκι πλέον για τον άνθρακα. Δεν υπάρχει μέλλον για τον άνθρακα. Και ε, αν θέλετε να την αγνοείτε αυτή την πραγματικότητα, συνεχίστε για χρόνια και χρόνια ακόμη να επιδοτείτε τα θρακοριχεία. Με πολύ βαρύ τίμημα. Πώς όμως μετά θα εξηγήσετε σε αυτούς οι οποίοι ε, πλήττονται, υποφέρουν από την κακή ποιότητα του αέρα, για το ότι... 400.000 ε, πρώιμοι θάνατοι στην Ευρώπη οφείλονται στα αναπνευστικά αυτά προβλήματα και δεν κάναμε τίποτα. Αυτό θέλουν ε, τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Νομίζετε θέλουν μια δουλειά στα θρακοριχεία. Όχι, άλλες δουλειές θέλουν. Και πιστεύω ότι με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα βρούμε και θα φέρουμε σε αυτές τις περιοχές ε, τις νέες θέσεις εργασία, ε, που δεν θα ασχολούνται πλέον με την εξόρυξη άνθρακα και δεν μπορούμε αυτή την προειδοποίηση, αυτό το μήνυμα να το αγνοούμε ε, και ούτε η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να το κάνει και ελπίζω ότι η Βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον θα συνεργαστούν χέρι-χέρι για να προχωρήσει αυτή η πράσινη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τίμερμανς και τώρα το λόγο έχει ο αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που καταδεικνύει ότι πραγματικά συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους. Συντοπίουμε ότι η κατάσταση είναι πήγουσα και θέλουμε όλοι να ευοδοθεί αυτή η ενεργειακή μετάβαση με τον τρόπο δίκαιο χωρίς αποκλεισμούς. Τούτων λεχθέντων θα πρέπει να συνεργαστούμε προς προς μία πράσινη και κοινωνικά βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας. Εμείς μπορούμε να δώσουμε μια κάποια καθοδήγηση, αλλά θα χρειαζόμαστε να έχουμε με το μέρος μας και τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε όμως την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε όλους τους απαραίτητους φορείς και όλους τους παράγοντες. Έχουμε τους κανόνες και έχουμε και την τεχνική υποστήριξη προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να έχουμε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια. Κατά αυτόν τον τρόπο τρόπο θίγω ορισμένα από τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε σήμερα, τα οποία έχουν να κάνουν με πολλές διαφορετικές πτυχές της ενεργειακής αυτής πράσινης μετάβασης, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι οι μελέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή καταδεικνύουν ότι θα έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία από τη μετάβαση αυτή προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα, σαφώς κάποιες θέσεις απασχόλησης θα εξαφανιστούν, όπως αυτές τις περιοχές που βασίζονται στον άνθρακα, αλλά θα δημιουργηθούν παράλληλα και νέες πράσινες θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζουμε τους πολίτες εκείνους και τις περιφέρειες εκείνες που θα θυγούν περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτό το μηχανισμό και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και αυτό ακριβώς πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημα αυτό το θέσατε πολλές φορές. Εμείς πραγματικά θέλουμε να έχουμε ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης με φρέσκο νοπό χρήμα πέρα και εκτός του υφιστάμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουμε το στόχο μας. Σας συνεργαστούμε λοιπόν προκειμένου ο στόχος αυτός να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτό το σημείο της Μερσιάς Διάταξης. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο, δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ε, είπα το της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για την κατάσταση στο Ιράν και το Ιράκ μετά την πρόσφατη κλιμάκωση. Να περιμένουμε μισό λεπτάκι να εγκατασταθεί ο κύριος Μπορέλ. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλώς ήλθατε, σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, συστηματική ανησυχία που δείχνει όσον αφορά την κατάσταση στις δύο αυτές χώρες που εμφανίζονται στο θέμα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα και που απασχολούν βέβαια και την ευρύτερη περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, η πρόσφατη κλιμάκωση τόσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση όσον αφορά την πρόοδο που είχαμε επιτύχει στην περιφέρεια αυτή τελευταία χρόνια και απειλεί τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Ξεκινώντας η συζήτηση αυτή, θα ήθελα να πω το εξή ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρο. Είπα εκπρόσωπος εκπρόσωπο και ω ε, αντιπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεσμεύομαι προκειμένου να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σταματήσει αυτό ο κύκλο βία στο Ιράκ. Πρέπει να σταματήσει αυτό ο κύκλο βία προτού τεθεί εκτό ελέγχου για μία ακόμα φορά. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο είμαι πεπισμένο ότι ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες οι οποίες ξεκίνησαν ήδη την προηγούμενη ε, Παρασκευή με το Συμβούλιο ε, Υπουργών Εξωτερικών, όπου μου δόθηκε εντολή να καταβάλω κάθε δυνατή διπλωματική προσπάθεια για να συμβάλλω στην αποκλιμάκωση τη όλη περιφέρεια, να συμβάλλω στον πολιτικό διάλογο και να προωθήσω μια περιφερειακή λύση ειρήνευση. Ακριβώ αυτά τα λόγια, αυτή τη διατύπωση βλέπουμε και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώ επίση και η πρόεδρος Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν συμβάλει σε αυτές τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και έτσι ακριβώ θα πρέπει να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι τελευταίε έξι εβδομάδε και ήδη από πέρυσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια, μια κλιμάκωση των εντάσεων στο Ιράκ που κορυφώθηκε με την εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμάνη από ένα αμερικανικό ντρόουν Είχαμε εν συνεχεία μία ανταπόκριση από το Ιράν και έπειτα ας μην ξεχνάμε ότι στις, στην ανταπόκριση αυτή, στα αντίπεινα του Ιράν, ευτυχώ δεν έχασε κανείς ε, την ζωή του, όσον αφορά δηλαδή τις αμερικανικές βάσεις που χτυπήθηκαν. Δεν θα πρέπει όμως να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εγώ ίδιος προσωπικά έχω αναλάβει δράση προκειμένου να οδηγηθούμε σε αυτοσυγκράτηση και σε αποκλιμάκωση από όλους τους παράγοντες εντός και εκτός της περιφέρειας, από το Ιράν ως το Ιράκ, από τις Ηνωμένε Πολιτείε στην Ρωσία, Ρωσία, την Κίνα και άλλους παράγοντες που εμπλέκονται. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι έχουν επιρροή στην περιφέρεια αυτή θα ασκήσουν επιρροή με τρόπο καλόβουλο, προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε την ένταση. Τώρα, για ποιο λόγο μα ανησυχεί τόσο πολύ η υφιστάμενη αυτή κρίση και πώ μπορεί η κρίση αυτή να επηρεάσει τα πράγματα και όλη την περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή στο Ιράκ βλέπουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Κατά αυτόν τον τρόπο δυστυχώ, θα αποδυναμωθούν όλε αυτέ οι προσπάθειε που γίνονται τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστεί το Ισλαμικό κράτο και οι μαχητέ του. Αυτό μπορεί να έχει πολλέ επικίνδυνε επιπτώσει. Ενδεχομένω οι μαχητέ του Ισλαμικού κράτου να αναλάβουν εκ νέου δράση και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση και ακόμα περισσότερου εκτοπισμένου από την περιφέρεια αυτή προ άλλε χώρε το κόστο θα είναι λοιπόν τεράστιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να διασφαλίσουμε τι σημαντικότερε επιτυχίε του παγκόσμιου συνασπισμού κατά του Νταέσσα. Η κατάσταση αυτή ενδεχομένως να μας αποπροσανατολίσει από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη αρχίσει να αναλαμβάνει το Ιράκ με την διαμόρφωση μια κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει και πάρα πολλέ οικονομικέ και κοινωνικέ προκλήσει, όπω την καταπολέμηση διαφθορά. Εμεί έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στη σταθερότητα και την οικοδόμηση του Ιράκ και έχουμε μια χρηματοδότηση η οποία περνάει τα 1,2 δισεκατομμύρια ήδη από το 2014 έχει εστιαστεί η χρηματοδότηση αυτή στην τροπιστική βοήθεια, στην υποστήριξη των εκτοπισμένων ανθρώπων, στην σταθεροποίηση περιοχών της χώρας που έχουν απελευθερωθεί, στη δημιουργία των απαραίτητων δυνάμεων ασφαλείας, όπως ακριβώς γίνεται και μέσω των συγκεκριμένων αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι με τη συνεχόμενη αυτή υποστήριξή μας, ότι οι μεταρρυθμίσεις που νόμιμα έχουν απαιτηθεί από τους Ιρακινούς πολίτες όντως θα ευοδοθούν και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι περαιτέρω δεσμεύσεις αναλήφθηκαν ήδη από το 2018 όσον αφορά την συνδιάσκεψη ανοικοδόμησης του Ιράκ που έγινε στο Κουβέιτ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ανταποκριθούμε και εμείς στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει με αυτά τα επιπλέον 400 εκατομμύρια τα οποία κινητοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να καταφέρουμε τελικά να προωθήσουμε τι οικονομικέ μεταρρυθμίσει κυβέρνηση και να δημιουργήσουμε βιώσιε με θέσει απασχόληση. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάσταση τώρα στο Ιράν είναι κάτι το οποίο εξακολουθούμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς. Είχαμε πολλά τραγικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα την συντριβή του αεροσκάφους των Ουκρανικών αερογραμμών, όπου 176 επιβαίνοντες χάσαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων πολλών πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριβή αυτή και όπως είπα και στην παρέμβασή μου στις 11 Ιανουαρίου πρόκειται για μια ιδιαίτερα θλιβερή τραγωδία και θα θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων και ελπίζω ότι το Ιράν θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί μας και ότι θα συνεχίσει να διεξάγει μια διαφανή έρευνα. Επίσης, την ίδια εβδομάδα 59 άτομα χάσαν τη ζωή τους καθότι ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελετών που γίνανε για την κηδεία του στρατηγού Σουλεϊμάνη και 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στις 9 Ιανουαρίου σε ένα τύχημα που είχε να κάνει με ένα λεωφορείο κοντά, στο, κοντά στην Τεχεράνη. Θα ήθελα να εκφράσω και στις περιπτώσεις αυτές πάλι τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο υφιστάμενο πλαίσιο έντασης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να προωθήσουμε την ασφάλεια και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην έχουμε περαιτέρω διάδοση των πυρηνικών όπλων. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τη συμφωνία αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Φαντάστε πώς θα ήταν σημερινή κατάσταση αν το Ιράν είχε και πυρηνικά όπλα. Και καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπήρχε το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόσφατα το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε στην πέμπτη κατά σειρά και τελική απόφασή του για να αναστείλει τους περιορισμούς που του έχουμε επιβάλει όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μα. ανησυχεί προφανώ η ανακοίνωση αυτή του Ιράν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να έχουμε κατά νου και τόσο μα λέει ο Διεθνή Οργανισμό Ατομική ενέργεια για το πώ θα εφαρμόσει το τελευταίο αυτό στάδιο άρση των περιορισμών το Ιράν. Ω συντονιστή του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράση, είμαι σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και με διπλωματικό τρόπο προσπαθώ πραγματικά να κρατήσω την ομάδα αυτή ενωμένη. Θα ακούσατε ενδεχομένω ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου της Γαλλίας και της Γερμανίας αναφέρθηκαν στο άρθρο 36, δηλαδή στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών που περιέχει το ε, κοινό αυτό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, θεώρησαν ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, να κινητοποιηθεί αυτό ο μηχανισμός επίλυση διαφορών, επειδή το Ιράν δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του κοινού ολοκληρωμένου σχέδιου δράσης. Ο μηχανισμός λοιπόν αυτό επίλυση διαφορών μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν θίξει Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Θα παρακολουθήσω λοιπόν εκ του σύνεγγυ αυτή τη διαδικασία και θα είμαι σε επαφή με όλου του συμμετέχοντε για τα επόμενα βήματα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω το εξή, ότι ο μηχανισμό επίλυση διαφορών είναι κυρίω μια διαδικασία προκειμένου να επιλύονται ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της συμφωνίας αυτή. Στόχος του μηχανισμού επίλυσης διαφορών είναι συνεπώς να καταφέρουμε να βρούμε μία λύση προκειμένου να επιστρέψουμε στην πλήρη συμμόρφωση στο πλαίσιο του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Δεν έχει να κάνει με την επιβολή κυρώσεων όπως ορισμένες εφημερίδες είπαν ήδη από σήμερα το πρωί. Όλοι οι συμμετέχοντες στη συμφωνία αυτή ήταν σαφείς ως προς την αποφασιστικότητά τους να διασφαλίσουν το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουμε την συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη. Χωρίς τη συμφωνία αυτή θα χάσουμε τελικά ένα πολύ καθοριστικό στοιχείο τη διεθνούς Αρτεκτονική για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και θα απολέσουμε τελικά ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό για τη διασφάλιση τη περιφερειακή ασφάλειας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουμε στην κλιμάκωση τη ένταση στην περιφέρεια αυτή. Κύριε Πρόεδρε, Πιέζει ο χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε δράση προκειμένου να επιλύσουμε την κρίση. Η ένταση στο Ιράκ καταδεικνύει ότι είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένη όλη αυτή η ευρύτερη περιφέρεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη Συρία μέχρι το Λίβανο, μέχρι την Ιεμένη αλλά και σε άλλε περιοχέ να καταφέρουμε να επιλύσουμε τα εφιστάμενα προβλήματα. Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή για το Ιράκ αλλά και για την ευρύτερη περιφέρεια, για το σύνολο του κόσμου τελικά και για εμά του ίδιου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ήδη υπάρχουν συγκεκριμένε εκκλήσει προ την Ευρώπη, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβει ένα, πιο σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι να συμβάλλουμε, όλοι μας, ενωμένοι ως ομάδα. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε κάποιε κρυφέ προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντικό οι εταίροι μας να εξακολουθούν να μας βλέπουν ως παράγοντα που θέλει να συμβάλλει στο διάλογο και στην επίλυση την ειρηνική όλων αυτών των διαφορών. Όπως στην αρχή της παρεμβασής μου, την προηγούμενη Παρασκευή, συγκάλεσα ένα έκτατο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη διάρκεια τη συνάντηση αυτής είπαμε εκ νέου ότι θα πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση. Επιβεβαιώσαμε επίσης ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ενότητα του Ιράκ, την εξαρτησία του Ιράκ και ότι θα πρέπει να έχει αδερφική εκαιρεότητα η χώρα αυτή. Και τονίσαμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με το Ιράκ και να συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε για την ανοικοδόμησή του. Τονίσαμε επίσης στα πλαίσια της συνεδρίασής μας αυτής ότι από κοινού είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι προ το συμφέρον μα να εξακολουθεί να ισχύει και προ το συμφέρον τη ευρύτερη περιφέρεια, αν θέλουμε να πετύχουμε πραγματικά ειρήνη και ασφάλεια και ήμασταν σαφείς στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής ότι θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση στην κρίση αυτή και ότι η λύση αυτή μπορεί να είναι μόνο περιφερειακή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε το ρόλο που μπορεί να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν έχοντας την υποστήριξη του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσωπικά θα συνεχίσω να, να ασχολούμαι με όλα αυτά τα ζητήματα, ερχόμενο σε επαφή, όπως σας είπα, με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, ταξιδεύοντας όπου αυτό είναι αναγκαίο και προσβλέπω ειλικρινά σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας προκειμένου να προωθήσουμε την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία της περιφέρειας αυτής που αυτή τη στιγμή τίθεται ένα αμφιβόλο εξαιτία των τελευταίων αυτών εξελίξεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Αντιπρόεδρε για την ε, πολύ πλήρη αυτή παρουσίαση της κατάστασης. Ξεκινά τώρα η συζήτηση. Θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Μίχαηλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστώ για την εισαγωγική σας παρέμβαση που τη συμμερίζομαι. Πράγματι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας ε, πιο ενεργός διαμεσολαβητής, ε, διότι ε, πράγματι υπήρξαν συνομιλίες και επαφές και με την Τεχεράνη. Καταφέραμε και εμείς να βοηθήσουμε στην αποκλιμάκωση ε, η Αμερικανή ε, Υπουργό ε, Άμυνα έκανε μια αντικειμενική δήλωση για την εκτέλεση του Σουλεϊμανή και είπε πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρα πολλά πράγματα. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως, δεν έχει λήξει αυτή η κατάσταση και πρέπει να ξέρουμε ότι τα κράτη της ε, μέλη, τα κράτη μέλη της ε, Ένωσης ε, πρέπει να κάνουν κάτι και έχουμε και τα, το, το Ιράκ που είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτη. Εσείς πρέπει να έχετε επαφή με το Ιράκ και πρέπει να βοηθήσουμε. Για το Ιράν τώρα Σίγουρα υπάρχει οργή με την κατάρρευση του ε, Ουκρανικού αεροσκάφους. Τρεις μέρες ε, γίνονται διαδηλώσεις ε, μετά την ομολογία. Ε, υπήρχαν ε, πάρα πολλοί που έχασαν τη ζωή τους. Ε, το θέμα είναι όμως ότι για να υπάρξει μετάνοια δεν αρκούν τα λόγια, αλλά θα πρέπει να υπάρξει η απόσυρση από το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις και ελπίζω με όλα αυτά να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο, η κάτι πήρε τώρα το λόγο. Κύριε Πατή, εκπρόσωπο. Για μία ακόμη φορά, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται πρωτοτελεσμένο γεγονότο. Η Αμερικανική κυβέρνηση και το Ιράν παίζουν με την παγκόσμια ασφάλεια. Και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίση αντιμετωπίζουμε πιθανό κίνδυνο ασφάλεια. Και η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλήμανι είναι η τελευταία μια σειρά προκλήσεων των Αμερικανών μετά την αποχώρησή του από, την από την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν. Και αυτό δημιούργησε ένα, ε, μια αλληλουχία ανασφάλεια στην περιοχή. Θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειε για να αποκλιμακώσουμε τα πράγματα και να διασώσουμε την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, όπως η ενεργοποίηση του μηχανισμού επίλυση διαφορών σήμερα. Ε, βέβαια, έχουμε διαφορετικά συμφέροντα από τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν αποσυρθεί από την περιοχή. Αυτό μόνο μπορεί να σημαίνει για μας. Ότι ήρθε η ώρα για μια ρεαλιστική συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας και την ασφάλειά μας. Φυσικά εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων του Ουκρανικού αεροσκάφου που συνετρίβει, που κατερρύφθη. Θα πρέπει οι Ιρανικέ αρχές να επιτρέψουν σε διεθνεί παρατηρητές να διεξαγάγουν διεξοδική και διαφανή έρευνα. Επίσης θα πρέπει το Ιράν να απόσχει από τη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών που κατέβηκαν στους δρόμου διαμαρτυρώμενοι για την κακή διαχείριση και τον αυταρχισμό του καθεστώτος. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να τάσεται υπέρ τη ενότητα και τη Δημοκρατία στο Ιράν και εν ανάγκη να εντείνει και την υποστήριξή τη προς τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Χίλντε Φάουτμαν. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς η ομιλήτρια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο τη δολοφονία του Σουλήμανη. Είναι πολύ πιο ευρύτερη. Και δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει εδώ. Οι Αμερικανοί θέλουν να αποχωρήσουν από τη Συρία, δολοφόνησαν τον Σουλήμανι και εμεί καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια ω απλοί παρατηρητέ και μαθαίνουμε από τι εφημερίδε και από τα ΜΜΕ τι προθέσει ε, των συμμάχων μα ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ καταρρίπτονται αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας και φυσικά νιώθουμε αποτροπιασμό δικαίως για μια τέτοια κατάσταση. Έχουμε δουλέψει σκληρά για την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν δεν θα πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Ευχαριστώ τον είπα το εκπρόσωπο για τη θέση που εξέφρασε και την άμεση δράση που ανέλαβε, αλλά δυστυχώς δεν αρκούν όλα αυτά. Το Ιράν κινδυνεύει να ξαναβυθιστεί στο χάος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσετε ώστε να συντονιστούμε και να έχουμε μια ενιαία φωνή και στάση στη Μέση Ανατολή. Δεν θέλουμε και πάλι για μια ακρόμη φορά να γίνουμε τα θύματα μιας μείζωνος μεταναστευτικής κρίσης. Είπατε ότι έχετε αναλάβει εντολή. Θέλω να σας δω σε αεροπλάνο, να πάτε στο Ιράν, να πάτε στη Washington και να διαβιβάσετε την ενιαία ευρωπαϊκή θέση για τα ζητήματα αυτά γιατί ξέρετε ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν ταυτίζονται ούτε με τα αμερικανικά ούτε με τα ρωσικά. Και αν κάποιος μπορεί να προασπίσει τα δικά μας ευρωπαϊκά συμφέροντα, αυτό είστε εσεί. Έχετε την απόλυτη υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έρνεστ Ουρτασούν. Ευχαριστώ. Κύριε Πατεκπρόσωπε, η αλήθεια είναι ότι οι αμερικανικές δράσεις και η δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανή παρολίγο να οδηγήσει σε χάος στην περιοχή, σε φοβερές ταραχές. Τώρα φαίνεται ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θέλει να σταματήσει κάτι που ήταν έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Είναι το μοναδικό που θα μας επιτρέψει μια ειρήνευση στην περιοχή και την αποφυγή μιας πυρηνικής κλιμάκωσης. Επίσης θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε με το Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χάρη σε αυτό το πλαίσιο που μας δίνει το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Είπατε ότι ενεργοποίησατε το μηχανισμό επίλυσης, επίλυσης διαφορών. Αυτό όμως ίσως ε, ερμηνευτεί διπλά. Μερικοί θέλουν να το φέρουν στο Σύμβουλο Ασφαλείας και να διατηρήσουν τη συμφωνία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ευκαιρία να συζητήσουμε παντός επιστητού. Να τηρήσει τις δεσμεύσεις του το Ιράν, αλλά να μιλήσουμε και για τις κυρώσεις που έχουν ε, επιβληθεί και πάλι και που κρατούν αχμάλωτα τη συμφωνία, συμφωνία πλήττοντας τον Ιρανικό λαό. Θα πρέπει με νύχα νύχια και με δόντια να τηρήσουμε και να υπερασπίσουμε αυτή τη συμφωνία, γιατί το διακύβευμα εδώ είναι η ασφάλεια των γειτονικών μας χωρών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διεθνή κοινότητα εύλογα ανησυχεί για την κλιμάκωση της έντασης στο Ιράκ και στην περιοχή μετά την επίθεση της Αμερικανικής, κατά της Αμερικανικής ε, πρεσβείας στο Ιράκ, ε, την δολοφονία του Σουλημανί και την κατάρριψη του Ουκρανικού αεροσκάφους ε, από Ιρανικό πύραυλο με 176 θύματα. Ε, δυστυχώς το Ιράν επηρεάζει και απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια γιατί ε, θα πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των πολιτών. Ε, δυστυχώς ε, δεν ε, ελήφθη υπόψη το μήνυμα της ΕΝΤΕ και το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήθελε να απαλλάξει από την ευθύνη του Ιράν. Ευτυχώς δεν ελήφθη υπόψη αυτή η έκκληση. Τρεις είναι οι άξονες της δημοκρατίας μας. ο σεβασμός της διαταφικής εκαιρεότητας των χωρών, η καταπολέμηση του σουνητικού ισητικού, ισλαμικού φονταματαλισμού και η προάσπιση των χριστιανικών μειονοτήτων στην περιοχή. Γιατί αυτές οι χριστιανικές κοινότητες είναι η πραγματική πολιτισμική γέφυρα μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Άννα Φωτίγκα. Σας ευχαριστώ. Κύριε είπατε εκπρόσωπε και Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα άλλο σημείο. Η, ε, η άρση της ε, ε δέσμευσης ε, των ε, λογαριασμών λόγω του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης δεν βελτίωσε την καθημερινότητα των Ιρανών. Συνεχίζεται η κλεπτοκρατία και η ευνοιοκρατία. Δυστυχώς είχαμε βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών. Έχουμε μεγάλη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, μεγάλη ανασφάλεια, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και τρομοκρατικών οργανώσεων και ανάπτυξη ε, βαλιστικών πυράβλων και των συναφών προγραμμάτων ανάπτυξης βαλιστικών πυράβλων. Για να μην μιλάμε για τις πρόσφατες ε, ε, δοκιμές πυράβλων μέσου βεληνικούς κατά βάσεων κατά του Ισλαμικού κράτους και την κατάρριψη του κρανικού αεροσκάφους πολιτικής αεροπορίας. Παρά τις εντάσεις αυτές, όπως και εσείς και εγώ ελπίζω να λάβει χώρα μια αποκλιμάκωση. Και η ενεργοποίηση του μηχανισμού επίλυσης των διαφορών είναι το ελάχιστο, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, εσείς και εμείς. Είναι το λιγότερο και ελπίζω ότι θα έχουμε και άλλους μηχανισμούς και εργαλεία στη φαρέτρα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κορνέλια Έρνστο. Είναι επόμενη. Ένα θέλω να πω. Και στις δύο χώρες ε, Έχουμε ε, ανθρώπους ε, που ε, διαδηλώνουν και φοβούνται και το νέο πόλεμο Απλά ε, αυτό που τους κάνει να διαδηλώνουν δεν είναι τόσο όλα αυτά όσο το ότι δεν αντέχουν άλλο. Έχουν πουχτήσει με την παρέμβαση της δύση ε, ε, και ουσιαστικά δεν τους επιτρέπουμε να καθορίζουν τη μοίρα τους με την απεικιοκρατία και όλα όσα έχουν ακολουθήσει και τα γνωρίζουμε με πολύ καλά. Πρώτα η Αμερική δεν είναι εφεύρεση του Ντόναλτ Τραμπ. Το ξέρουμε εδώ και καιρό. Ε, και δεν έχουμε ακούσει τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις δύο χώρες. Πρέπει να τους σεβαστούμε ε, και δεν θα πρέπει ε, ουσιαστικά μετά από πολιτικές δολοφονίες να χύνουμε κροκοδίλα δάκλια ή να στέλνουμε κάποιες, κάποια συλληπιτήρια και μιλάμε για την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων γιατί αυτό θα, που θέλει το Ιράκ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία της χώρας αυτό είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα ολοκληρώνεται αυτό ο γύρος με τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Καταδικάζουμε την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ με θύματα μεταξύ άλλων Ιρανούς και Ιρακινούς στρατιωτικούς. Καταγγέλουμε το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να κηρυχθεί Ανατολή επικράτεια του ΝΑΤΟ η επικίνδυνη εμπλοκή της ευρωπαϊκής ένωσης στο πλαίσιο κλιμάκωσης των ανταγωνισμών για έλεγχο της ενέργειας στόχο έχει να επωφεληθεί η ίδια. επικαλείται τα ίδια προκλητικά προσχήματα δικαιολόγησης πολέμων όπως στη ιουγκοσλαβία στη συρία στο ιράκ στη λιβύη στο αφγανιστάν που καταδικάζουν τους λαούς σε προσφυγιά και δυστυχία. εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας με το ουκρανικό αεροπλάνο για την οποία έχει τεράστια ευθύνη η ιρανική κυβέρνηση τονίζουμε ότι η απροκάλυπτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην πολιτική των ηνωμένων πολιτειών και η διαχρονική τεράστια ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν μετατρέψει την ελλάδα σε αμερικανονοτοϊκό στρατόπεδο θέτουν τον ελληνικό λαό σε μεγάλο κίνδυνο. να ενταθεί λοιπόν η λαϊκή πάλη για να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία Ελλάδα ηνωμένων πολιτειών για να κλείσει τώρα η βάση της ούδας και όλες οι βάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ενημερώσω όσους έχουν ζητήσει το λόγο ότι από εδώ και πέρα όλοι όσοι πάρτε το λόγο θα έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Δεν, το, ε, δεν θα το επαναλάβω στον καθένα. Η κυρία Σκίτενταλ, να έχετε υπόψη σας. Ο καθένας έχετε ένα λεπτό από εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Ο Κασέμ Σουλεϊμανή ήταν από κάθε άποψη τρομοκράτης. Και ναι, δεν νομίζω κανένας από εμάς εδώ στην Ολομέλη να θρυνεί το θάνατό του. Βέβαια, δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη τη συνέπειες αυτού του χτυπήματος και οι εξελίξεις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα μας δείξουν την πορεία που θα ακολουθήσει αυτή η ευάλωτη περιοχή και ιδιαίτερα στο μέλλον. Επίση, ε, ε, διαδηλωτέ έχουν συλλέψει του δρόμου του Ιράν και του Ιράκ, Βαγδάτη, Τεχεράνη, ε, κατά του αυταρχικού καθεστώτο και θέλουν να αποφασίσουν για το πεπρωμένο τους πέρα από ξένε παρεμβάσει. Το Ιράκ είναι η χώρα που περισσότερο επηρεάζεται από την Ιρανική παρεμβολή στα εσωτερικά του. Χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανάκτηση κυριαρχίας και τη σταθερότητά του. Γι' αυτό θα ήθελα κύριε Μπορέλ να μας πείτε με λεπτομέρειες ε, ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες σας στο μέλλον για το Ιράκ και με ποιο τρόπο η ΑΕΔ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, είπα για τα λόγια του Συμφωνούμε απόλυτα τόσο εγώ προσωπικά όσο και η ομάδα μας. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μείωση της έντασης στην περιοχή. Η δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμάνη είχε πολύ χειρότερες συνέπειες, ε, μάλλον θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερες συνέπειες αυτές που είχε, Και πρέπει να δούμε αν θα πετύχει η Ευρώπη αυτά τα οποία επιδιώκει στο πλαίσιο τη Δετής Πυρηνική Συμφωνία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μα. Και αυτό ο μηχανισμό ε, Instex ε, για την ε, συναλλαγή με το Ιράν. Επίσης έχουμε την, το μηχανισμό επίλυσης αντιπαραθέσεων που κινητοποιείται και αυτό είναι λογικό γιατί το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι δεν θα τηρήσει τις ρήτρες συμφωνίας και δεν το έχει κάνει ήδη και κατά το παρελθόν. Έχει επίσης δολοφονήσει διαδηλωτές ε, και στο Ιράκ, στο Λίβανο, στη Σύρια και στην Ιεμένη. Ουσιαστικά στηρίζει ε, τις ε, ομάδες εκεί, ε, το Ιράν και αυτά όλα πρέπει να πάψουν. Ευχαριστώ πολύ, Χόργουερτ. Ευχαριστήσω τον κύριο Μπορέλ για την παρέμβασή του και να τον ευχαριστήσω για τα ειλικρινή συλληπιτήριά του που εξέφρασε για όλες αυτές τις ζωές που έχουν χαθεί και στα πλαίσια βέβαια της πτήσης των Ουκρανικών αερογραμμών. Σαφώς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βασιζόμαστε στη διπλωματία και όχι στις απειλές και τις προσβολές στο Twitter. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έτυχε κάποιες διαβούλευσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ας μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ποια ήταν η στάση και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την υφιστάμενη κυβέρνηση όσον αφορά τη στάση που διατηρεί απέναντι στην πολιτική του Τραμπ για την όλη αυτή περιφέρεια. Νομίζω ότι ο δικός μας ο Πρωθυπουργό ζήτησε να αντικατασταθεί αυτή τη στιγμή η συμφωνία που έχουμε με το Ιράν με μια συμφωνία την οποία θα προωθήσει ο πρόεδρος Τραμπ και εξακολουθεί παράλληλα να λέει η ε, κυβέρνηση του Μένου Βασιλείου ότι θέλει να προωθήσει τη συμφωνία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω εμεί να προωθήσουμε τη δική μα συμφωνία και να συνειδητοποιήσουν άλλοι, όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να, εκφράζονται όλε οι απόψει και στα πλαίσια του Ιράν και του Ιράκ χωρί να υπάρχει ο φόβο των αντιπίνων. Ευχαριστώ. Νόημαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό επίλυση των διαφορών για να διασώσει τη συμφωνία με το Ιράν. Και επίση να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα, να γίνουμε διαμεσολαβητέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και άλλων τοπικών ε, παραγόντων για να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Αυτό έχει αναφερθεί ήδη. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο σημαντικό. Η δολοφονία του Σελιμανί πιθανόν να επισκιάσει ε, τις φωνές των διαδηλωτών που ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις εδώ και μήνες και στο Ιράν και στο Ιράκ. Από την Παρασκευή όμως ε, ε, ξανακατέβηκαν στους δρόμους αυτοί οι διαδηλωτές παρά τις απειλές και είναι ακόμη πιο ηχηρή η φωνή τους. Θα ήθελα λοιπόν δράση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει αυτού του διαδηλωτέ από τη βία και τι ε, δολοφονίε. Να καλύψουμε το κενό που θα αφήσει η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιοχή και να στείλουμε με διπλωματικό τρόπο ένα σαφέ μήνυμα στο καθεστώς του Ιράν. Φυσικά ε, θα είμαστε ε, η πολιτική της ήπιας δύναμης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε ειρήνη στην περιοχή, αν και πάλι ε, φημωθούν ή σιωπήσουν οι διαδηλωτές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την προλαλή σας καταρχήν γιατί είπε πολλά σοβαρά πράγματα που αληθεύουν και όλα. Και σίγουρα το ιρανικό καθεστώς είναι αυταρχικό και πολύ Ισλαμικό τα τελευταία 40 χρόνια και εδώ και χρόνια διαπραγματευόμαστε με το Ιράν για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου, τι αρχέ και τι αξίε μα. Αλλά όπω βλέπουμε δεν είχαμε και μεγάλη επιτυχία. Και τώρα, αν οι Αμερικανοί δολοφόνησαν έναν υψηλά ιστάμενο του Ιράν, έναν στρατηγό που ήταν τρομοκράτης και οφείλεται και ευθυνόταν για τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ιράκ, το Λίβανο, στη Συρία. Τώρα πολλοί Ευρωπαίοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους και λένε αυτό είναι παράδεκτο, θα πρέπει να τιμωρήσουμε τους Αμερικανούς γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση αυτή οι Αμερικανοί είναι οι σύμμαχοί μας. Και υπάρχει και ένα απλούστατο ερώτημα. Θα στηρίξουμε τους Αμερικανούς, θα σταθούμε στο πλευρό τους για να ε, επιτύχουμε τη σταθερότητα γιατί ε, ακριβώς υπήρχε επιτυχία τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του φόβου των Ιρανών ε, για τους Αμερικανούς. Θα πρέπει λοιπόν αυτούς να υποστηρίξουμε, τους Αμερικανούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια ερώτηση με τη διαδικασία της μπλε κάρτας, αγαπητέ συνάδελφε. Τη δέχεστε? Βεβαίως. Ο κύριος Κούλογλου. Κύριε ε, Μάντισον, όταν δεν έχουμε εμπόλεμη σύραξη, η δολοφονία ενός υψηλού αξιωματούχου μιας χώρας από άλλη χώρα αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Είστε υπέρ του σεβασμού και της στήρισης του διεθνούς δικαίου, ναι ή όχι. Ο κύριος Μαρίζων. Συμφωνώ με την ερμηνεία σας του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν είναι κατά του διεθνούς δικαίου η ε, θανάτωση ενός τρομερού τρομοκράτη. Αυτό δεν είναι... Η δεν είναι κατά του διεθνού δικαίου. Γιατί ευθύνεται για πολλέ τρομοκρατικέ επιθέσει, ευθυνόταν αυτό ο άνθρωπο. Και οι Ιρανοί πολλέ φορέ δήλωσαν ότι δεν έφεραν ευθύνη για τι ε, επιθέσει. Οπότε, αν μιλήσω εγώ για το ε, διεθνέ δίκαιο, θα ήθελα να πω ότι οι Αμερικανοί ακριβώ το αμερικανικό δίκαιο, το διεθνέ δίκαιο εφάρμοσαν. Προστάτευσαν τη χώρα του ε, από από εξουδετερώνοντας αυτόν τον επικίνδυνο τρομοκράτη. Ευχαριστώ Κύριε Κάνκο. Σας ευχαριστώ. Η κρίση στο Ιράν είναι η πρώτη δοκιμή της νέας γεωπολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι συμφωνούμε από ό,τι φαίνεται ότι ο στρατηγός Σουλεϊμανή που έχασε τη ζωή του έχασε τη ζωή του μετά από μία δράση βίαιη, μετά από όλες αυτές τις βιοπραγίες που είδαμε τελευταία χρόνια εξαιτία του. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μας να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά ζήτησε να υπάρξει μία αποκλιμάκωση και δυστυχώ, 176 άνθρωποι ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους άμεσα εξαιτία τη κλιμάκωση τη κατάστασης. Νομίζω ότι ε, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λυγίσουμε μπροστά στον Ιρανικό εκφοβισμό. Θα πρέπει να καταφέρουμε να ξανασφέρουμε το Ιράν πίσω στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με το Ιράκ προκειμένου να περισσώσουμε τον παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ντάεσ. Βρεθήκαμε στο χείλο πάλι του πολέμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναφέρουμε όλα τα μέρη γύρω από το τραπέζι του διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης ήταν ιδιαίτερα καθοριστικό. Ο κύριο Γουάλλα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να δολοφονήσουν παράνομα τον στρατηγό Σουλημανή καθώς επίσης και πολλούς άλλους εξωματούχους, καταδεικνύει το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο πιο αποσταθεροποιητικός και επικίνδυνος παράγοντας στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε διεξάγουν ένα πόλεμο κατά τη τρομοκρατία, ενώ οι ίδιε τρομοκρατούν, οι ίδιε ρίχνουν βόμβε, οι ίδιε αποσταθεροποιούν. Του ζητήθηκε να αποχωρήσουν από το Ιράκ, αλλά θα αποχωρήσουν τελικά από το Ιράκ, θα αναγνωρίσουν τη δημοκρατική αυτή απόφαση που έλαβε το Κοινοβούλιο του Ιράκ, θα σεβαστούν πραγματικά το δίκαιο της χώρας. Κύριε Επίτροπε, δεν συμφωνείτε κι εσείς ότι η περιφέρεια αυτή με όλους αυτούς τους παράγοντες τελικά είναι πολύ πιο ασφαλής με την απουσία των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι οι πρώτε οι οποίε δεν εφάρμοσαν το πυρηνικό αυτό, την πυρηνική αυτή συμφωνία. Και ποιο είναι ο ρόλο επίση του Ισραήλ. Για ποιο, το, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται αυτή τη στιγμή να υποστηρίζει την τρομοκρατική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Καστάλντο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το νέο αυτό έτος ξεκίνησε πολύ γρήγορα με μια νέα κρίση. Η απόφαση του Πενταγώνου να δολοφονήσει τον Κασέμ Σουλεϊμανί, νούμερο 2 στο Ιράν μετά τον Αλή Χομενεή, αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην ακολουθεί το διεθνές δίκαιο, καθότι μάλιστα έγινε και σε ένα τρίτο κράτος, στην επικράτεια του Ιράκ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ακολουθείται μια εντελώ λανθασμένη στρατηγική από τι ΗΠΑ, μια στρατηγική που βασίζεται μόνο στη δύναμη, στην ισχύ, στη βία και βία που εξυπηρετεί μόνο, τα αμερικανικά συμφέροντα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε όταν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή επιβάλλονται τόσο βίες οικονομικές κυρώσεις εκ νέου κατά του Ιράν. Εμείς νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό με έναν τρόπο θετικό ε, ερχόμενοι σε επαφή με τρόπο διπλωματικό με τον Υπουργό ε, Τζαβάτ Σαρίφ, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μαζί του να διευρύνουμε ή δυνατόν ακόμα περισσότερο το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, προκειμένου αυτό πραγματικά να ελοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σικόρσκι. Κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δικαίω εξουδετερώσαν τον ε, στρατηγό Σουλεϊμάνη που ήταν ένας ε, ξεδιάντροπος οργανωτής τρόμου τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Και ε, το Ιράν είναι μια χώρα που ταυτόχρονα αποτελεί και την αιτία της εξάπλωσης ε, της τρίτης ουτοπίας ε, του 21ου αιώνα, τη θεοκρατία δηλαδή. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε με το Ιράν. Γιατί ενώ μερικές φορές ε, έχουμε σχέσεις με το καθεστώς, η ίδια η φύση του καθεστώτος εμποδίζει το Ιράν να γίνει ένας φυσιολογικός και υπεύθυνος εταίρος οι Ιρανοί και πάλι κατέβηκαν στους δρόμους ε, και διαμαρτύρονται, γιατί θέλουν να ζουν σε μια φυσιολογική χώρα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του βοηθήσουμε, αλλά να μην υπερβάλλουμε κιόλα, γιατί λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για αυτού για τον Ιρανικό λαό, ιδιαίτερα όταν δρούμε εθνικά. Ε, το θέμα αυτό έχει πολλά διακυβεύματα και ε, βραχυπρόθεσμα ίσως έχει περισχύσει ο Τραμπ, αλλά θέλουμε ενωμένη νέα προσέγγιση του συνόλου της Ευρώπης ε, και ε, αμέριστη υποστήριξη των δράσεών σας, κύριε είπατε, εκπρόσωπε από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σβέν Μίξερ. Τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε το Ιράν ε, και τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, να έχουν μια κλιμάκωση των σχέσεων που κορυφώθηκε με τη δολοφονία του Σουλεϊμανί και την κατάρριψη του κρανικού αεροσκάφους. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι ήταν καταστροφικός ο ρόλος του Σουλήμανη στην περιοχή και είχε στα χέρια του το αίμα πολλών αθώων ανθρώπων. Πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ε, πλήρως εμπλεκόμενες Ηνωμένες Πολιτείες στο διεθνές προσκήνιο. Πιστεύω βέβαια ότι είναι κρίσιμη σημασία ε, ο τρόπος που ασκεί το παγκόσμιο του ρόλο ο Ηνωμένες Πολιτείες να είναι υπεύθυνο. Και όταν ε, αναλαμβάνει δράσεις που έχουν τόσο μνημειώδεις συνέπειες, οι δράσεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν τμήμα μιας συνολικής και ρεαλιστικής στρατηγικής, για να μην δημιουργηθεί ένα, μια, ένα που θα διαφύγει το ελέγχου μας ε, και μια αποκλιμάτωση έντασης που θα οδηγήσει σε χάος στην περιοχή. Αυτό είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να μην φυστούμε προσπαθειών για να αποκλιμακώσουμε αυτή την έκρηθμη κατάσταση και να εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον ύπατο εκπρόσωπο προκειμένου να ε, πορευθεί προς αυτό το στόχο και να κρατήσει ζωντανό το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Λουαζό. Εδώ και δεκαετίες ε, το Ιράν βρίσκεται στο κέντρο της, της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Αλλά η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα και δεν μπορούμε να δούμε τελικά πώς θα βγούμε από την κρίση. Απέναντι στο Ιρανικό αυτό καθεστώς, το οποίο ασχολείται περισσότερο με την επιβίωσή του, ποιο θα είναι το τίμημα. Η αμερικανική πολιτική τη μέγιστη πίεση δεν έχει κάνει την περιοχή αυτή πιο ασφαλή. Βλέπουμε ότι δεν ακολουθείται αυτή τη στιγμή η συμφωνία τη Βιέννη. Βλέπουμε ότι υπάρχει με ακλιμάκωση στην ευρύτερη περιφέρεια. Βλέπουμε ότι ο Λίβανο βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να ακουστεί η φωνή τη Ευρώπη, η φωνή τη λογική. Α επαναλάβουμε τι προτεραιότητέ μα. Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καταπολέμηση του Ντάεσ οι προτεραιότητε αυτέ μα βρίσκουν όλου σύμφωνου, έτσι δεν είναι. Επομένω, θα πρέπει να λάβουμε δράση και α μην παραμένουμε αδρανεί απέναντι στην αποθήκη που έχουμε στην άμεση γειτονία μα. Βασιζόμαστε στη δική σα δράση, κύριε Αντιπρόεδρε. Η κυρία Ροέτη έχει το λόγο. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, όπω είπα Αριστοτέλη, μπορούμε να δεχθούμε κατηγορίες μόνο για αυτά τα οποία εξαρτώνται από εμά. Τι εξαρτάται όμως από εμά αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση στο Ιράν πραγματικά μας κάνει να ασχοληθούμε με το όλο πάζλ της Μέσης Ανατολής. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η Ουκρανία είναι παράπλευρο θύμα της όλης αυτής κρίση. Πώς μπορούμε όμω να μην υποστηρίξουμε τους πολίτες του Ιράν που στρέφονται κατά του καθεστώτος, κατά των στρατιωτών της χώρας αυτής που ρίξανε το αεροπλάνο αυτό. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει εδώ πέρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην καταλήξουμε σε αυτό το ανθρώπινο λάθος, όπως είπε το Ιρανικό καθεστώς. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Θα πρέπει να επιρρύψουμε ευθύνε εκεί όπου πραγματικά έχουμε άσκηση βία από κάποιον που ήταν ε, ο σύμμαχός μας. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να επιρρύψουμε την ευθύνη σε αυτόν ο οποίο προκάλεσε την κλιμάκωση και όχι σε αυτού οι οποίοι μέσω αντιπίνων προσπαθούν να απαντήσουν. Ο κύριο Μαριανή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια για το ε, Ιρανικό καθεστώ που ανετράπει το 2003 ούτε και για το σημερινό, αλλά η Δύση είναι σαφέ ότι φέρει μεγάλη ευθύνη στο χάος ε, που με την υποστήριξη πολλών των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών φέρουν οι ΙΠΑ, να τρέπονται το καθεστώς του 2003 και ε, διαδίδοντας ψευδείς ειδήσει που είναι σήμερα της μόδας ε, ως έκφραση. Η καταγγελία επίσης τη πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν, ενώ δεν έδειχνε τίποτα ότι δεν τη σέβονται, ήταν κάτι που οδήγησε σε μια νέα περίοδο ασάφειας και για μια ακόμη φορά η Ευρώπη είναι ανίκανη να διεξαγάγει ανεξάρτητη πολιτική. Πώ να ζητήσουμε το Ιράν να τηρήσει τη συμφωνία τη Βιέννη ενώ ε, υφίσταται ακόμη κυρώσει και ιδίω τις πληρώνει ο λαό. Αν θέλουμε αποκλιμάκωση πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να έχει συναλλαγέ με τη χώρα παρακάμπτοντας τις κυρώσει. Ε, θα πρέπει να γίνει σεβαστή η ψήφο ε, του Ιρακινού Κοινοβουλίου για τα Αμερικανικά στρατέματα να αποχωρήσουν. Αυτό το οποίο έχουμε καταστήσει σε αυτή τη χώρα σπήραμε ε, θύλε και θερίζουμε τρομοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε τις διαμαρτυρίες των Ιρανών κατά της δικτατορίας, του καθεστώτος που δολοφονεί αμάχους και επίσης ε, και στο Ιράν είχαμε παλιά ε, διαδηλώσεις κατά της δικτατορίας του Σάχη. Αλλά και το καθεστώς των Αγιατολάχ ε, θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο της περιοχής και δημιουργεί προβλήματα στην Τεχεράνη. Ο στρατηγός Σουλήμανη ήταν από τους ε, προτεργάτες αυτής της πολιτικής του Ιράν. Θα πρέπει τώρα να αφήσουμε κατά μέρους ε, τη πολιτική της κυρίας Μογκερίνη. Θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο Ιράν. Ο κύριος Μπαρένα Άρσα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η πολιτική δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί εκ μέρου των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε ένα σπιράλ βία όχι μόνο στο Ιράν και το Ιράκ, αλλά σε όλη την περιοχή και ήταν ίσω το σημείο εκκίνηση ενό νέου είδου ψυχρού πολέμου ή πολέμων δια την προσώπου που κάποιε ε, παγκόσμιες δυνάμεις είναι διατεθειμένε ε, να παίξουν στην περιοχή. Θέλουμε να παρατηρήσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να διευκολύνουν το διάλογο και την οικονομική ανάκαμψη περιοχή με πρόγραμμα αρρωγή και να μην ενδώσουμε σε κλήσει για το εμπάργκο που ιστορικά χρησιμεύσε μόνο για να τιμωρήσει του πιο ανήμπορου ε, και ε, ανυπεράσπιστους κοινωνικούς ε, κλάδους, τους πιο εύθραυστους πολίτες του Ιράν και του Ιράκ. Επίση θα πρέπει ε, να, αποσυ... να αποχωρήσουν τα ξένα στρατεύματα όπως ζήτησε το Ιράκ, το στρατεύμα των ΗΠΑ και να τηρηθεί η διεθνής νομιμότητα που παραβιάστηκε με τη δολοφονία του Σουλιμανί. Επίσης, ε, όλη η επαναφορά στην ε, ε, κανονικότητα θα πρέπει να γίνει χωρίς εξωτερικές παρεμβολές, κάτι που προϋποθέτει εξάλληψη κάθε μορφής παρεμβατισμού, είτε αυτός προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε την ερώτηση με μπλε κάρτα από την κυρία Πεχουμέα Πεχουμέα. Βεβαίως. Κυρία Μπεχουμέα Μπεχουμέα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαρένα καταδικάστηκε το 2016 από το δικαστήριο για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ που δολοφόνησε πάνω από 800 Ισπανούς πολίτες και ακόμη 300 εγκλήματα δεν έχουν διελευκανθεί. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Μπαρένα εσείς κύριε Μπαρένα καταδικάζετε ή όχι την τρομοκρατία του ΕΤΑ. Γιατί αν καταδικάζετε τη βία του ΕΤΑ, στην οποία πρωταγωνιστήσετε κι εσείς, ε, θα ήθελα να το ακούσω από το στόμα σας. Καταδικάζετε την τρομοκρατία. Ο κύριος Μπαρένα είναι ε, μέλος ε, του Μπίλντου, του κόμματος που επέτρεψε το σχηματισμό κυβέρνησης από τον Πέντρο Σάντσες και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπαρένα για μισό λεπτό. Κυρία Μπεχουμέα, ε, Ακούγοντά σα, διαπιστώνω ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στη χώρα το Βάσκο τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν υπάρχει πια έτα, δεν υπάρχει πολιτική βία, τουλάχιστον εκ μέρου των Βάσκων. Και κλείνει αυτό ο κύκλο με την αναγνώριση των θυμάτων και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Κυρία Μπεχουμέα, η θέση σα πόρο απέχει από την συνεννόηση και την επανασυμφιλίωση. Και μάλιστα το κόμμα σα ακόμη φαίνεται ότι υιοθετεί μια στάση εκδίκηση ε, θα ήθελα να στεριστείτε και εσείς τη διαδικασία ε, της ειρήνευσης και της πολιτικής συμφιλίωσης που εδραιώνεται στο σύνολο της βασικής κοινωνίας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριο Σίντσιτς. Τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και το Ιράκ δείχνουν την αλαζονία και την υπεροψία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ε, και μάλιστα είναι η υπεροψία και έπαρση να δολοφονούν ε, πολίτη, στρατηγό μάλιστα ε, άλλης χώρας, στο έδαφος της χώρας αυτής, είναι ε, υπεροπτικό να χάνεται αθώοι πολίτες και να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ε, είναι επικίνδυνη η στρατηγική του κυρίου Πομπέο, του Υπουργού Εξωτερικών και μάλιστα θα πρέπει προσπαθεί πάση θυσία να αποφύγει την ε, συζήτηση στο Κογκρέσο. Σίγουρα η αξιοπιστία δεν είναι το δυνατό σημείο ε, της αμερικανικής πολιτικής. Θυμάστε τα μέσα μαζικού ολέθρου ε, και τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Μπούς. Και το αποκορύφωμα της υπεροψίας είναι να πει κανείς ότι